Mesdames, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες σήμερα. Οπότε, παρακαλώ ελέγξτε ότι έχετε την κάρτα ψηφοφοριών σας. Και θα αρχίσουμε ευθύς αμέσως την ψηφοφορία του σχεδίου ψηφίσματος, ενδιαμέσου ψηφίσματος, των Μπέγκιο και Κάλφιν. Οι εισηγητές και οι συνεργάτες μας εργάστηκαν μέχρι και βαθιά στη νύχτα για να διατυπώσουν συμβαστικές τροπολογίες. Καθίστε παρακαλώ, έχετε τους καταλόγους ψηφοφοριών. Υπάρχει ένα ειδικό φυλάδιο με ψηφοφορίες. Ένας κατάλογος ψηφοφοριών. Οι εισηγητές έχουν ε, πληροφορίες ή επεξηγήσεις. Όχι, όχι, ωραία. Οπότε, συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην παράγραφο 2, προφορική τροπολογία των εισηγητών, υπενθυμίζοντας την σημασία υγιών δημοσίων οικονομικών υπέρ. Κατά ε, ε κυρία Ανδρέασεν, υπενθυμίζοντας τη σημασία των υγιών ε, δημοσιονομικών είναι δικό σας θέμα. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 της Γκουε υπέρ. Η Γκουε κατά. Οι υπόλοιποι. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 Ashworth. Εισηγητής κατά. Α, καταπίπτει. 24 τη Συντόνια. Συγητές υπέρ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 του Σαλβαδόρ, εισηγητές υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 των εισηγητών, υπέρ, κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτουν οι επόμενες 32 της ΕΛΓΑ. Οι εισηγητές είναι κατά υπέρ. Η πράσινη κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. Επόμενη παράγραφος 33. Μάρτα Ανδρέασεν. Οι εισηγητές κατά υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34. Αντζουνταφ. Με μια προφορική τροπολογία των εισηγητών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 Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57. Οι εισηγητές είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58. Οι εισηγητές είναι κατά. Υπέρ. 3. Κατά. Η πλειοψηφία απορρίπτεται. 59 της ΓΚΟΕ. Οι εισηγητές κατά. Υπέρ. Οι εισηγητές είναι κατά. Είναι μια πληροφορία που σας δίνω, δεν είναι σύσταση. Υπέρ, υπέρ, και πράσινη, κατά. Οι υπόλοιποι αποχές απορρίπτεται. Οπότε, η 60. Η 60. Της Έλγα, οι είναι κατά, υπέρ. κατά τα μαμούθ. Αποχές απορρίπτεται. 61 συντόνια. Η σύγητας είναι κατά υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας της συντόνια. Βεβαίως η συντόνια. 3, 4 κατά αποχές απορρίπτεται. 62 της Γκουε. Οι εισηγητές είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 των εισηγητών. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά πρέπει να ψηφίσουμε την 63 της ΓΚΟΕ που αποδέχονται οι εισηγητές αν είναι προσθήκη. Α, όχι, με συγχωρείτε. Α, με συγχωρείτε προτείνει η Γκουε μία προσθήκη, την οποία δεν θέλουν οι συγητές, εντάξει, ποιοι είναι υπέρ. Γκουε πράσινη, κατά, υπόλοιποι, αποχές, απορρίπτεται. Εγκρίνεται λοιπόν η συμβαστική 7 χωρίς αυτή την προσθήκη. Συμβαστική 8 των εισηγητών, υπέρ. Κατά, ένας κατά αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην 74. Οντί. Οι κατά. Υπέρ. Η Κατά. Οι υπόλοιποι. Αποχέ. Απορρίπτεται. 75. Χαουγ Και Φερνάντες. Οι είναι υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 76. Καρβάλιο. Οι είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 των εισηγητών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 των εισηγητών υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Το ΕΛΚ έχει όντως ζητήσει κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα με ε, κέντρο προσοχής στις, πιο, στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Α, ναι. Όλο το κείμενο εκτός αυτές τις λέξεις, χωρίς τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά δύο. Αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα, αυτές τις λέξεις, με τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά Λοιπόν, πρέπει να ε, ελέγξουμε. Οι συγητές είναι υπέρ της προσθήκης αυτής. Οι συγητές είναι υπέρ. Υπέρ, υπέρ, βεβαίως. Είναι περίπλοκο. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Λήξη. 22 υπέρ 12 κατά, δύο αποχές. Εγκρίνεται αυτή η προσθήκη. Λοιπόν, με κέντρο της προσοχής ε, η, της λιγότερο από τις περιοχές. Και αυτό θα συμπεριληφθεί. Εντάξει. Όλον τον υπόλοιπο συμβασμό, λέει ο πρόεδρος. Α, τον έχουμε ήδη ψηφίσει. Μάλιστα, βεβαίως. Ωραία. 90 του Σαλβαδόρ έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές, τρεις κατά αποχές, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε μία μικρή τροπολογία της Γιούτα, την 103. Οι συγκητές είναι υπέρ, υπέρ, κατά άποχες, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 των εισηγητών με την τροπολογία, την προφορική τροπολογία. Α, πρώτα θα ψηφίσουμε την... Μισό λεπτό. Ο κύριος εισηγητής. Μπέγκε. Πρώτα τη συμβαστική 12 και μετά την προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Ωραία, πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. Συμβαστική 12 χωρί την προφορική υπέρ. Κατά αποχές. Η προφορική τροπολογία να αντικαταστήσουμε τα προγράμματα για την νεολαία με το πρόγραμμα εγγύηση για την νεολαία. Ποιοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κάποιοι από το ΕΛΚ είναι κατά, αλλά περισσότεροι είναι υπέρ. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. 5. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Των συγκριτών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111. Νταφ. Συμβατός προσθήκη. Αλλά οι συγητές είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 των εισηγητών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μια μικρή προσθήκη 121 τη Συντόνια. Οι εισηγητέ είναι κατά. Υπέρ. Δύο. Κατά. Υπόλοιποι. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 των εισηγητών. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124. Οντί οι εισηγητέ είναι κατά. Υπέρ. Κανείς. Οπότε βεβαίως απορρίπτεται. 125. Τη συντόνια εισήγητες είναι κατά. Υπέρ. Η συντόνια. Η κυρία, η πράσινη και η γκουε. Κατά. Οι υπόλοιποι αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε 126-127 του Ρίτσορντ. Ναι. Όχι. η Γκουε κάνει διαφοροποιήσει ε, στι ε, τροπολογίε τη άκρα δεξιά, τέλο πάντων. 126. Οι συγκητές είναι κατά υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. 127. Υπέρ. Η Γκουε είναι υπέρ. θα το αρέσει του Ρίτσο. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 128 του Άιντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 Τη συντόνια εισηγητές κατά υπέρ 4 κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 18 των εισηγητών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 19 των εισηγητών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την 133 της Έστερ Ντελάνια ως προστίκη. Οι εισηγητές είναι κατά, υπέρ. Τρεις, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Έχει εγκριθεί 19 χωρίς την τροπολογία 133. Συμβαστική 20 έχοντας υπόψη ότι η 137 θα ήταν προστίκη. Θα ψηφίσουμε μετά. Καλά. Η συμβαστική 20 χωρίς την 137, έτσι. Εφόσον μας λέει ο Ξαβιό ότι είναι σωστό, φανεί, ξέρεις. Υπέρ κατά αποχές. Ωραία. Τώρα την 137 ως προσθήκη. Οι συγκητές είναι κατά. Υπέρ. Οκτώ. Κατά. Πάνω από από Αποχές απορρίπτεται. 142-143. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Όχι. Όχι. Καλά. 142. Άσουερ. Εισηγητές κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143. Υπέρ. 3. Κατά. Αποχές απορρίπτεται επίσης. 144. Πίπα. Οι είναι υπέρ. υπέρ. Κατά. 7 αποχές εγκρίνεται 145 πίπερ αλλά οι είναι κατά υπέρ 2 α με συγχωρείτε με συγχωρείτε 4 κατά αποχές απορρίπτεται 146 ντελάνγκε οι είναι κατά υπέρ Κανείς δεν υποστηρίζει την Έστερ. Πάει. 148 Ashworth υπέρ. Κανείς υπέρ του Ρίτσαρτ. Πάει και αυτή. 149 της Χέλγα με την προφορική τροπολογία που είναι υπέρ. Οι υπέρ. Κατά. τρει αποχές εγκρίνεται με την ε, προφορική προστίκη. 150 είναι συμβατή, αλλά οι συγητές είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. 4 κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151 του Ρίτσο. Οι κατά. Υπέρ. Η Γκουε κατά. Οι υπόλοιποι αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην 152 του κλούτε. Οι συγκεκριτές είναι κατά. Υπέρ. 3. Κατά. 4 υπέρ. Μάλιστα κατά αποχές απορρίπτεται. 153-154 μαζί. Α, ωραία, ευχαριστώ Άλτα. Οι συγκεκριτές είναι κατά υπέρ. 1 κατά αποχές απορρίπτονται. 155 Ανδρέασεν. Οι συγητές είναι κατά υπέρ. Ένας κατά. Οι περισσότεροι. Αποχές απορρίπτονται. Οπότε 156 με την προφορική προσθήκη των εισηγητών ούτω ώστε να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα οι θεσμοί ε, ε, υπέρ. Κατά ένας κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο κατά μάλιστα. Ο κύριος Φέρμ. Ένα σχόλιο για τις επόμενες δύο τροπολογίες. Είναι για το θέμα της ε, ενιαίας έδρας. Υπάρχει πολύ μικρή διαφορά, αλλά θα πρότεινα μεταξύ αυτών των δύο τροπολογιών, δηλαδή θα προτείνω όσοι είναι υπέρ ενιαίας έδρας να απορρίψουν την πρώτη τροπολογία του Άσουερθ, όχι για την εκακή, αλλά γιατί 158 είναι ακριβώς η διατύπωση που έχουμε στην έκθεση Σούλερ και νομίζω ότι θα πρέπει να εμείνουμε να μην συγχύσουμε την κατάσταση με τη διαφορετική διατύπωση που προτείνει ο Άσχουερτ. Προτείνω λοιπόν να καταψηφίσετε την 157 και να υπερψηφίσετε την 158. Ευχαριστώ. Ωραία, λέει ο πρόεδρο. Ο Ρίτσαρντ δεν είναι εδώ, δεν μπορούμε να του στήσουμε λοιπόν από την τροπολογία του. Ωραία. 157. Οι συγητές είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 του Γκόραν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 των εισηγητών. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην, στην 162 συντόνια με προφορική ε, ε, τροπολογία να απαλληφθεί που θα ε, ε, επηρεάσει τα ποσά που είναι ήδη προκαθορισμένα ούτως ώστε όχι να υπέρ κατά τρεις αποχές εγκρίνεται. 163, ο που είναι συμβατή, αλλά οι συγητές δεν τη θέλουν υπέρ. Κανείς δεν είναι με τον άρα εξαφανίζεται. 164, ο D, οι συγητές δεν θέλουν υπέρ. Κανείς, κανείς, καλά. Πάει και αυτή. 165-166 μπορούμε να τις πάρουμε μαζί. Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Του Ρίτσορντ, οι συγητές είναι κατά υπέρ. Ένας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική 23. Των εισηγητών. Θα ψηφίσουμε το προφορικό τμήμα μετά. Ωραία, την προφορική τροπολογία. 23 χωρίς την προφορική τροπολογία της Άλντε. Υπέρ. Κατά. Ένας κατά. Εγκρίνεται. Η προφορική τροπολογία να, να προσθέσουμε η αυστηρή εφαρμογή του κανόνα ε, N συν 2 για όλα τα κράτη-μέλη χωρίς εξαιρέσεις. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται χωρίς αυτήν την προφορική τροπολογία η συμβαστική 23. 168. Μίλντερ. Οι είναι υπέρ. Υπέρ κατά κανείς. Αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 48 έχουμε μία προφορική τροπολογία των εισηγητών χωρίς τις λέξεις η συνέχιση του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 169 έχει αποσυρθεί. 170 του Ρίτσορντ εισηγητές είναι κατά υπέρ. είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. 171 της Γκουέ. Δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα οι εισηγητές είναι υπέρ. Ποιοι άλλοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνει. Το δεύτερο τμήμα οι εισηγητές είναι κατά υπέρ Κατά οι υπόλοιποι αποχές το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 172 Νταρντέν με μια προφορική τροπολογία των εισηγητών. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 των εισηγητών υπέρ κατά ένας κατά αποχές εγκρίνεται. 175 του Γκέραν οι συγητές είναι υπέρ, υπέρ. Κατά ένας κατά αποχές εγκρίνεται. 176. Α, ναι, ναι, βεβαίως. 176. Τη Συντόνια. Συγητές είναι κατά. υπέρ ποιοι είναι παρακαλώ. Ένας. Μία. Μία. Μία μισή. Όχι, μία. Δύο. Α, δύο. Κατά αποχές απορρίπτεται 177 της Άλντα οι είναι κατά υπέρ Ιγκουέ κατά υπόλοιποι αποχές απορρίπτεται 178 του Άντζου Νταφ με την προφορική τροπολογία των εισηγητών. Υπέρ ποιοι είναι παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 179 Άιντερ ρησίτες είναι υπέρ, κα, υπέρ λοιπόν κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε μαζί 180 και 181 της Γκουε ωραία οι εισηγητές είναι κατά υπέρ η Γκουε και η Πράσινη κατά οι υπόλοιποι πάνω κάτω αποχές απορρίπτονται συμβαστική 25 υπέρ κατά Δύο. Αποχές Δύο. Εγκρίνεται. 186. Άλντα. Οι συγκεκριτές είναι κατά. Υπέρ. Η Γκουε. Και ένας πράσινος. Α, ούτε καν. Ούτε καν. Η Γκουε. Μάλιστα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 187. Τη Συντόνια. Οι συγκεκριτές υπέρ. Υπέρ. Κατά ένας. Αποχές. Εγκρίνεται. 188 ευρώ. Του Λάσλο έχει αποσυρθεί 189. Του George Lyon. Εισηγητές κατά. Υπέρ. Ένας. Δύο, τρεις. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 190 ντάφ εισηγητές είναι. Κατά υπέρ Κανείς υπέρ του Άντριου. Εξαερώνεται. 191. Συντόνια. Υπέρ. 2. 3. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 192 του Άντζου. Οι συγητές είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. 3. Αποχές. Εγκρίνεται. 193 του Ρίτσορντ εισήτες. Είναι κατά, υπέρ. Κανείς. Εξαφανίζεται. 194 έχει αποσυλθεί. 195 του Ρίτσορντ. Εισηγητές κατά, υπέρ. Ένας. Αποχές. Απορρίπτεται. 196. Τη συντόνια. Οι θέλουν Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα μέχρι εκεί που λέει ώστε να το πιο σύντομα. Οι εισηγητές είναι υπέρ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, όπως κάθε καθυστέρηση και τα λοιπά, οι εισηγητές είναι κατά υπέρ, δύο, κατά αποχές, το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Δεν έχει έρθει ακόμα καφές. Όχι ακόμη. Ο καφές έρχεται μόνο άμα ψηφίσουμε ένα ορισμένο αριθμό τροπολογιών. Α, Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ωραία. Άλτα. Τις 197-198 μπορούμε μαζί. Ωραία εισηγητές κατά, υπέρ. Ουδείς αποχές, κατά αποχές, απορρίπτονται 199, συντόνια, εισηγητής κατά, υπέρ. Τέσσερις υπέρ, έως και πέντε, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμό 25 των εισηγητών, υπέρ. Κατά ένας. Αποχές εγκρίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ψηφίσουμε τις ε, επόμενες. Τι νόημα έχει ο συμβασμός. Τέλος πάντων, 200 εισηγητών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 201 του Ρίτσαρτ. Εισηγητές κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ουδής. Απορρίπτεται. 202. Νταφ. συγητέ κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ουδής. Ε, υπερασπίζεται το Νταφ. Καταστράφηκε. Αιτιολογικές σκέψεις. 3. Ρίτσαρτ. συγητέ υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Της Χέλγκα που είναι συμβατή. συγητές υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ κατά. Ένας αποχές εγκρίνεται. πέντε. Ρίτσαρντ. Εισηγητές υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. πέντε. Ε, έξι βλέπω. Αποχές εγκρίνεται. Με διαφορετική πλειοψηφία. σύνδυασμός 26 των εισηγητών υπέρ. Κατά. Ένας. Αποχές εγκρίνεται. 9 της Χέλγκα εισηγητές κατά. Ποιοι είναι υπέρ. 4. 5. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 της Χέλγκα εισηγητές είναι υπέρ αυτή τη φορά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 της Χέλγκα με μια προφορική των εισηγητών για την ε, απαλυφή του πολίτη. Καλυπέρ. Κατά. Δύο. Αποχές. Βγαίνει η λέξη political. Εγκρίνεται. 12 της Χέλγκα. Οι εισηγητές είναι κατά. Ποιοι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 27 των εισηγητών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16. Νταφ. Οι συγητέ είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ του Άντρου. Ένα. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Αιτιολογικέ σκέψεις. ένα Γιάν Μούλτερ. Με μία προφορική των εισηγητών υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 2. Ζαν Πιεροντή οι συγητές κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Η γκουε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Το κείμενο στο σύνολό του. Α, λεπτό. Le vote final, donc le vote est ouvert. Άρχεται η συνεδρίαση, ε, η συνεδρίαση, με συγχωρείτε, η ψηφοφορία. 40 κάρτες, 37 πρέπει να ψηφίσουν, τρεις κοιμούνται, παρά τον καφέ κοιμούνται, οι τρεις. Πέρας, δεν ψήφισαν οι τρεις τελούν εν υπνώση. 34 υπέρ, 1 κατά, 2 αποχές. Να συγχαρούμε τον εισηγητή. Εξαιρετική εργασία. Γνωρίζετε τι ψηφίσατε. Θα ήθελα όμως να πω στους υπολείπους, τους παρόντες, ότι εγκρίναμε μία, ένα συμβιβασμό, μία τροπολογία συμβιβασμού που λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση των άλλων επιτροπών. Ε, δυνάμει της παραγράφου 66 τονίζει τη σημασία των ε, γνωμοδοτήσεων των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίζουν κατευθυντήρες γραμμές για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπως ορίζεται από αυτό το ψήφισμα. Θεωρούμε ότι οι συστάσεις θα πρέπει να τροφοδοτήσουν τα αντίστοιχα πολιετή προγράμματα. Επίσης θεωρούμε ότι η ειδική νομοθετική διαδικασία του MFF, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με θέματα που αφορούν την ε, τακτική νομοθετική διαδικασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιθυμούσε η ομάδα επαφής υπό την προεδρία του Σούλτς. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε αρχίσει αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο και το ίδιο θα ακολουθήσουμε να κάνουμε εάν εγκριθεί αυτή η διαδικασία από την Ολομέλεια. 11 Οκτωβρίου σήμερα η διαδικασία διαπραγμάτευσης είχε αρχίσει πέρσι στις 12 Οκτωβρίου, αλλά στην ουσία οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν σε μερικές μέρες. Λοιπόν, δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε με το πολιετές, γιατί έχουμε και την έκθεση του Jean-Luc Dean. Έχετε τον κατάλογό σας για την έκθεση του Jean-Luc. Ως προς τον κανονισμό, που αφορά τον φόρο προσθέμενες αξίες. Έχουμε τέσσερις τροπολογίες της Ιζαμπέλ Ντουρόν, οι συγητές, οι υπέρ μπορούμε να τις ψηφίσουμε μπλοκ. Ωραία. Επί των τεσσάρων της Ντυράν. 1, 2, 3, 4 υπέρ. Κατά. Ένας. Αποχές. Εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 5. 5 και 6. Της Ιζαμπέλ Ντουιράν. Από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 7 του Ρούμπιχ έχει αποσυρθεί. Άρα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την έκθεση του Ζαν Λουκ. Αρχίζει η ψηφοφορία. 39 κάρτες έχουμε πλέον. Α, 40. Αλλά ψήφισαν μόνο 36. Άρα τι κάνετε, βάζετε τις κάρτες σας για να μην ψηφίσετε, δεν σας καταλαβαίνω. 37-38. Α, βλέπω ότι συνεχίζεται παρά τη λήξη. 35 υπέρ, ένας κατά, δύο αποχές. Να συγχαρούμε τον Ζαν Λουκ για την εξαιρετική του εργασία. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Όμως, όμως, είχαμε συμφωνήσει χτες μετά από αίτημα της Ίγκε Γκρέσλε και αίτημα του Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες ότι θα ασχοληθούμε με τη μεταφορά 3, μεταφορά πίστοσης που αφορά την ΕΙΕΔ και θα υποβάλαμε το ερώτημα αυτό σε εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ. Με βάση το ερώτημα του εισηγητή και της Ίγκε Γκρέσλε. Ο κύριος Τιχερή Μπουσέ είναι παρόν, εκπρόσωπος της ΕΙΕΔ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό ως προς τις διοικητικές δαπάνες. Θέλει να μιλήσει καταρχήν ο εισηγητής, μετά η Ίγκε. Όπως επιθυμείτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπα εχθές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτά που προελέχθησαν εν μέρη. Μιλάμε για μία μεταφορά πίστοσης προς πληροφόρηση, δηλαδή μιλάμε για μία μεταφορά ενός 10%. Θα ήθελα όμως να κάνω μία σύσταση για τις επόμενες μεταφορές να υπάρχει σαφήνεια και αυτό το τονίζω στην ΕΙΕΔ, γιατί αυτό το καθεστώς θα πρέπει να διέπει τις μεταφορές πιστώσεων. Βλέπουμε ότι η ΕΙΔΕΔ έχει αρχίσει να λειτουργεί σχετικά πρόσφατα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να ψηφίσουμε αυτή τη μεταφορά πίστες, παρόλο που δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια. Βάση περιπτώσει, επειδή είναι μόνο για πληροφόρηση, μπορούμε να το κάνουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τη συνάδελφό μου κατά πόσο θέλει κάτι να προσθέσει και γι' αυτό ζητήσαμε και διευκρινής από τον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Συμφώνω με την Ίγκες σε αυτά που είπε χθε και ελπίζω να μην έχουμε νέα προβλήματα στο μέλλον. Υπενθυμίζω, λέει ο Πρόεδρος, ότι πρόκειται για μια μεταφορά που σχετίζεται με θέματα της ΕΙΕΔ που μας υποβλήθηκε προς πληροφόρηση. Η Ίγκε Γκρέσλε όμως έθιξε μία σειρά ζητημάτων χτες και της δίνω το λόγο έτσι ώστε ο κύριος Μπουσέ να μας απαντήσει. Ίγκε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Η μεταφορά πιστώσεων τροποποιεί τον προϋπολογισμό που αποφασίσαμε. Είναι υποχρέωσή μας να υποβάλλονται αυτά τα αιτήματα με τρόπο που να έχουμε ε, πλήρη πληροφόρηση για το τι αλλαγή προκαλεί αυτή η μεταφορά πιστώσεων στον προπολογισμό. Με βάση την ε, πρόταση της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης δεν είναι σαφές ποια ποσά θα πάνε από κεφάλαιο σε κεφάλαιο ή και από τίτλο σε τίτλο. Οπότε η παρουσίαση μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος, γιατί μπορεί να θεωρήσουμε λοιπόν ότι μεταφέρονται 4,5 εκατομμύρια, αλλά εάν υπολογίσουμε επακριβώς με τον υπολογιστή στο χέρι, με το κομπιτεράκι, είναι πολύ περισσότερα. Θα ήθελα λοιπόν να μπορέσουμε να επανέλθουμε για το θέμα αυτό, ούτω ώστε να δούμε ποιο ποσό πάει από πού, πού γιατί αλλιώ έχουμε περίεργα αποτελέσματα. Στη γραμμή 3.000 μισθή υπαλλήλων σε αντιπροσωπείες η αιτιολόγηση είναι τέτοια που δεν αιτιολογεί τα ποσά διότι με αυτόν τον τρόπο ενώ λέγεται ότι υπάρχει ένα ε, έλλειμμα 6,4 εκατομμυρίων, λέγεται ότι θα δημιουργηθούν 23 νέες θέσεις. Δεν το κρίνω αυτό, δεν επικρίνω τη δημιουργία των 23 νέων θέσεων, αλλά υπολογίζεται ότι για 9 μήνες είναι 280.000 ευρώ το ποσό για μια θέση. Αυτό είναι υπερβολικά μεγάλο ποσό, διότι Ε, ε, με άλλους υπολογισμούς ε, λέγεται ότι είναι 370.000 το κόστος μιας τέτοιας δημιουργίας θέσης για αυτό το ποσό. Άρα υπάρχουν με πολλές ανακρίβειες. Πραγματικά είναι παραπλανητικό και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Παρακαλώ τον κύριο Μπουσέ να κάνει τις αιτήσει του όπως τα άλλα θεσμικά όργανα ήμουν σε επιτροπές που είδαμε μεταφορές πιστώσεων, αιτήσεις μεταφορών πιστώσεων από άλλα θεσμικά όργανα που είναι πολύ λογικότερες και πολύ καλύτερα διατυπωμένες και σας, ευχαριστώ. και σας παρακαλώ πολύ να το κάνετε και εσείς με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε. Ίγκε, ο κύριος Μπουσέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οπωσδήποτε θα βελτιώσουμε την κατάσταση για την επόμενη φορά ως προς τις ε, μεταφορές ανατίτλο, όπως ζήτησε η κυρία Γκρέσλε. Μιλάμε για μία μεταφορά 4,5 εκατομμυρίων ως προς την έδρα της αντιπροσωπείας και θα τονίσουμε, θα σταθούμε στις αντιπροσωπείες. Ζητήσαμε 20 θέσεις ΑΝΤΕ για το 2012 και μία θέση ΑΝΤΕ για τις αντιπροσωπείες 2012. Και πρόκειται για 4,5 εκατομμύρια συνολικά, δηλαδή τόσα θα εξοικονομήσουμε. Μιλάμε για 14 εκατομμύρια 409.000, 31.000 ευρώ του τίτλου 1 και 32 περίπου εκατομμύρια στον τίτλο 2. Ε, για να βάλουμε 4 εκατομμύρια περίπου στον τίτλο 3. Ως προς τους μισθούς αντιπροσωπείες είχαμε μία πρόβλεψη δαπανών για το 12 και ο μόνος τρόπος είναι να ξεκινήσουμε από τα ποσά που καταβλήθηκαν το Σεπτέμβριο του 12 που είναι που τα βλέπετε στον πίνακα και είχαμε ορισμένες δυσκολίες γιατί έχουμε 20 νέες θέσεις με πιστώσεις που ισχύουν από τα τέλη Οκτωβρίου. Όταν προσλάβαμε το 12 έπρεπε να τους πληρώσουμε να καταβάλουμε μισθούς για 12 μήνες. Δηλαδή μιλάμε για ένα 1% του προϋπολογισμού. Θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο προϋπολογισμός του 2013 και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να καταβληθούν οι μισθοί για το επόμενο έτος. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι προσλήψεις. Έχουν αρχίσει, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί. Μιλάμε περίπου για 88 εκατομμύρια περίπου. Και μιλάμε για 104 εκατομμύρια συνολικά, αν λάβουμε υπόψη και τα επιδόματα. Σε σχέση με το 12 έχουμε περισσότερους υπαλλήλους τους οποίους ε, πληρώνουμε από ό,τι είχαμε προβλέψει κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο στις αρχές του 2011. Τότε δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά η οποία είναι και μοναδική. Αυτή η διαφορά δεν αφορά νέες θέσεις, απλώς έχουν καταληφθεί οι προϋπάρχουσες θέσεις που είναι υψηλότερες από τις προεβλεπόμενες σε σχέση με το 2012 ως προς το 2013. Και μιλάμε για ένα δίκτυ 5,1%. Αυτή είναι η διαφορά. αν έρχεται σε ένα 5,1% σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. και έχει το λόγο. Με συγχωρείτε, αλλά δεν διευκρινίστηκε η κατάσταση, πρέπει να πω. Ε. Δεν έγινε σαφέστερη η κατάσταση. Δεν μπορείτε παρακαλώ να το κάνετε όπως όλοι οι άλλοι ούτω ώστε να κάτσω στο γραφείο μου και να μπορέσω να κοιτάξω τα στοιχεία στο γραφείο μου με ησυχία, να μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνατε. Δεν θέλω να σας δημιουργήσω δυσχέρειες. Θέλω να υπάρξει διαφάνεια. Αυτό είναι η πρώτη μου αίτηση. Να έρθω σε αυτά που είπατε για την πλήρωση των θέσεων. Με βάση αυτά που είπατε, γράφετε από 498 θέσεις εάν ε, λέτε ότι θέλετε ότι θέλετε να δημιουργήσετε 23 καινούριε. Ε, ε, αν διαρρέσω το 6,4 για το 32 φτάνω σε 370.000. Είναι πολύ ακριβό αυτό. Ακόμη και αν ξέρω ότι είναι ακριβή πάλι. Και τι άλλο υπάρχει. Τι άλλο υπάρχει. Μετά είπατε ένα ποσοστό 5,1 και 8,45. Ποσοστά. Υπέθεσα ότι αυτά τα ποσοστά είναι αντανάκλαση των ε, αριθμών, των αριθμητικών στοιχείων. Δεν καταλαβαίνω. Ε, αναφέρονται και σε άλλα στοιχεία αυτά, άλλες 20 θέσεις. Θέλω απλώς να μου πείτε γιατί κοστίζει τόσο πολύ αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλώ γραπτός, γραπτός. Μα με συγχωρείτε δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Βέβαια είμαι περιορισμένος να το αλλά δεν το κατάλαβα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Ίγκε για τις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστούμε κύριε Μπουσέ για τις απαντήσεις σας. Αλλά τις χρειαζόμαστε και γραπτός. Εδώ δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε τη διαχείριση της ΙΕΔ, αλλά θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση και αυτό είναι φυσικό. Η ΙΕΔ είναι ένα νέο όργανο της Ένωσης, μια νέα υπηρεσία Κατανοούμε ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα όσο σιγά σιγά αρχίζει να λειτουργεί και να διαχειρίζεται εσωτερικά και να, εφαρμόζεται, να εφαρμόζει τον κανονισμό της. Από ό,τι είπε ο κύριος Μπουσέ, εγώ κατάλαβα ότι ένας λόγος της μεταφοράς αυτής είναι όχι μεν ότι αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων κατά τη χρήση του προπολισμού αλλά για το ότι τη στιγμή που πληρώθηκαν θέσεις δεν ήταν ακριβώς όσες και αυτές προβλέπονταν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε χρειαζόμαστε όλες τις αποσαφηνήσεις και πληροφορίες γραπτός και όσο το δυνατόν το συντομότερα. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν τελειώνει και αυτό το σημείο και περνάμε τώρα στο 8 δηλαδή την έκθεση του Ρίτσαρντ Άσουρθ για το πρόγραμμα Ηρακλής 3. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μάλιστα, Ηρακλής 3. Τον Δεκέμβριο του 2011 η Κομισιόν ενέκρινε μια πρόταση κανονισμού για το Ηρακλής 3 για την προώθηση δράσεως στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Αυτό το νέο πρόγραμμα τονίζει ιδιαίτερα την καταπολέμηση του παθητικού καπνίσματος αλλά και του ενεργητικού και της λαθρεμπορίας σιγαρέτων. σύμφωνα με πληροφορίες που αφορούν τέσσερις διεθνείς εταιρείες καπνοβιομηχανίες. Φυσικά όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στα συμφέροντα, στα διάφορα συμφέροντα που υπάρχουν μέσα στην ε, Ένωση, αλλά υπάρχει και το διοικητικό κόστος της λειτουργίας του προγράμματος και οι επιπτώσεις του στον προϋπολογισμό, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του πολιετούς πλαισίου στην πρόταση αυτή πρέπει να αποφευχθούν οι επικαλύψεις μεταξύ κομισιών και κρατών μελών με τα δικά τους αντικαπνιστικά και αντιαπατικά προγράμματα. Και το λένε αυτό οι τροπολογίες ιδιαίτερα οι δύο. Επίσης πρέπει να βρούμε συνέργειες και με άλλους οργανισμούς και προγράμματα ώστε να μειωθεί το κόστος του προγράμματος και να διασφαλιστεί τελικά η προστασία των φορολογουμένων. Πρέπει πρώτα να δούμε τα αποτελέσματα ανεξαρτήτων μελετών. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ηρακλής 2 ήταν επιτυχής. Γι' αυτό διαγράφω την τελική πρόταση της τροπολογίας 3. Επίσης δέχομαι την ε, έκθεση του ε, ελεγκτικού συνεδρίου σχετικός, αλλά νομίζω ότι έπρεπε προηγουμένως να είχαμε τύχη διαβούλευσης για να να είχαν τύχη διαβούλευσης από τους ενδιαφερόμενους για να, και τα κράτη-μέλη για να ληφθεί υπόψη. Γενικά υποστηρίζω την ε, αξιολόγηση του ελεγκτικού συνεδρίου, ιδιαίτερα την ανάγκη να είναι οι σχετικές μελέτες ανεξάρτητες και να λαμβάνουν υπόψη τους πλήρως την φοροστιθέμενη ενωσιακή αξία που θα είχαν τέτοια προγράμματα. Δηλαδή να συγκριθούν τα αποτελέσματα με τους προτινόμενους στόχους και να ληφθούν μαθήματα για τα μελλοντικά προγράμματα όπως και μέχρι το 20. Αυτή είναι η λογική των τροπολογιών μου 4, 5, 6 και 7. Σημερίζομαι και άλλα μια της έκθεσης των ελεγκτών πιστεύω ότι ο ανώτατος ρυθμός συγχρηματοδότησης πρέπει να μην ξεπερνάει το 50% αλλά παρόλα αυτά συμφωνώ επίσης ότι σε εξαιρετικέ και δεδικαιολογημένες περιπτώσεις πρέπει να μπορεί να αυξάνεται η συγχρηματοδότηση μέχρι το 80%. Και αυτό το λέω στην τροπολογία 12. Όσο για τη γενική χρηματοδότηση της εφαρμογής του προγράμματος για την περίοδο 14 με 20 είναι 110 εκατομμύρια. Πράγμα το οποίο αποτελεί σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τον Ηρακλή 2. Και σε αυτά τα πλαίσια και μέσα στο γενικότερο πολιετές πλαίσιο θα ζητούσα λιγότερα, μικρότερα ποσά. Να δούμε δηλαδή σε ποιους τομείς μπορούμε να πετύχουμε εξοικονομήσεις και στις τροπολογίες 8, 9 και 10. Αυτό ακριβώς λέω. Ελπίζω να μπορέσουμε επικοδομητικά να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε μία σωστή γνωμοδότηση και προσμένω τα σχόλια των άλλων εισηγητών και συναδέλφων. Ευχαριστούμε Ρίτσαρντ. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Δεν είμαι ισκιώδης αλλά θα ήθελα να πω ορισμένα θέματα γιατί είναι σημαντικό αλλά και λυπηρό συγκρούσεως μεταξύ της Ένωσης και κρατών μέλων στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Επανειλημμένα έχουμε τσακωθεί και με την Όλαφ που δικεί το πρόγραμμα αυτό για τα θέματα αυτά. Διαπιστώνουμε πλήρη αδιαφάνεια για το πώς ε, αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό Γι' αυτό, Ρίτσορτ, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες όπου θέλουμε να υπάρξει παρακολούθηση. Τι γίνονται με τα χρήματα, τι γίνονται τα χρήματα αυτά. Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί έκαναν κάποιες ε, επιφυλάξεις, ε, διατύπωσαν επιφυλάξεις. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται. Θέλουμε για πρώτη φορά από τότε που υπάρχει το πρόγραμμα αυτό μια έκθεση για το πώς αξιοποιούνται οι πιστώσεις. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα μεγάλα κονσέρν της ε, καπνοβιομηχανίας ε, κατέθεσαν 2 δισεκατομμύρια για να καταπολεμηθεί ε, το λαθρεμπόριο, αλλά κατά 90% τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στους εθνικούς προπολογισμούς και από αυτό το 10% που μένει στον κοινοτικό προπολογισμό πρέπει να συγχρηματοδοτήσουμε επενδύσεις στα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σιγαρέτων. Καταλαβαίνω αυτά που μας λέτε, αλλά η Όλαφ θα ήθελε να ανέβει η συγχρηματοδότηση στο 80%. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον 80% και τα κράτη μέλη 20%. Οπότε το θέμα είναι από πλευρά δικαιοσύνη. Δεν είναι σωστό αυτό. Και τα χρήματα ούτως ή άλλως που έχουν πάρει τα κράτη-μέλη εδώ και πολύ καιρό τα έχουν δαπανίσει. Έχουν ε, λοιπόν δαπανηθεί τα χρήματα αυτά και δεν υπάρχει καμία υποδομή για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. ούτε, ούτε καν στα κράτη της Βαλτικής που είναι η θύρα εισαγωγής για το λαθρεμπόριο. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τον τρόπο υποβολής εκθέσεων, το reporting, να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται κάθε χρόνο με τα χρήματα που δαπανούμε, ιδίω για την ε, υποδομή. Θέλουμε μια υποδομή που να δημιουργηθεί και επιπλέον να λειτουργεί σε μερικά χρόνια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτή την υποδομή, τι έχει γίνει, τι πρέπει να γίνει ακόμη. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτή ως Επιτροπή Προϋπολογισμών να επηρεάσουμε αυτό το θέμα που είναι σημαντικό και για την Ένωση και για τα κράτη-μέλη της. Ο κύριος Γκάια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημερίζομαι αυτά περί πολιτικής ε, δικαιοσύνης που είπαν οι Άσουέθ και Γκρέσλε εφόσον είναι κοινό μας καθήκον με βάση το άρθρο 25 ε, προστασία των οικονομικών σφαιρών της Ένωσης το, απλή, το απλούστερο θα ήταν 50% να πληρώνουν τα κράτη-μέλη και 50% η Ένωση. Έτσι δεν είναι. Ωστόσο, η Ένωση και ο πλανήτης είναι κάπως πιο περίπλοκος από ένα τέτοιο απλό συλλογισμό. Από τις εκθέσεις της ε, Europol ξέρουμε πώς πάνε οι ροές ε, παραχαραγμένων και ε, λαθρέων προϊόντων. Υπάρχουν ε, διάφοροι δρόμοι και μέσω Ιταλίας και μέσω των Βρετανικών νησιών και εκείνοι που θίγονται κυρίως είναι η Αυστρία. Έχουν κάποια αεροδρόμια μόνο. Εκεί είναι πιο απλά λοιπόν για την Αυστρία, αλλά για άλλες χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα, η Αυστρία δεν έχει, είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Απειλούνται πολύ περισσότερο. Για παράδειγμα, για την Ελλάδα ξέρουμε το κράτος, όπως ξέρετε στην Ελλάδα, ε, δεν είναι και τόσο πρόθυμο να κάνει δαπάνες για το θέμα αυτό. Αλλά πρέπει να χρηματοδοτήσει παρόλα αυτά αυτά τα προγράμματα από τα στοιχεία που έχουμε ενώπιόν μας για τις ζημίες που προκαλούνται. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο το κόστος από τα 10 δισεκατομμύρια, είναι 10 δισεκατομμύρια, 9 για τα κράτη-μέλη και 1 για τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό. Όπως ξέρουμε λοιπόν, κάθε ευρώ που ε, επενδύεται για αυτό το πρόγραμμα μας προστατεύει ιδιαίτερος εφόσον δυσχεραίνει το λαθρεμπόριο και σημαίνει ότι έχουμε περισσότερα έσοδα και περισσότερους ίδιους πόρους ως Ένωση. Αλλά εφόσον ε, θίγονται διαφορετικά τα κράτη-μέλη και έχουν διαφορετικά καθήκοντα, συμμερίζομαι την πρόταση της ίνια ότι πρέπει να μας υποβάλλονται εκθέσεις ούτω ώστε να καταλαβαίνουμε ποια χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί για ποια ε, μέσα. Ξέρετε ότι χρειαζόμαστε πολύ ε, προηγμένα τεχνολογικά μέσα. Ξέρετε ότι τα περνάνε τα ε, λαθρέα τσιγάρα μέσα σε τεράστια φορτηγά, οπότε είναι πολύ σοβαρό από τα διάφορα λιμάνια που περνάνε στο Ρότερνταμ και τα λοιπά να μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και πρέπει να ξέρουμε πώς γίνονται αυτά. Πρέπει να δούμε ποιος είναι καλύτερα να το κάνει αυτό, τα κράτη-μέλη, η Ένωση, τι προσωπικό πρέπει να αξιοποιήσουμε, πώς πρέπει να το εκπαιδεύσουμε κτλ. Θα πρέπει, όπως είπε και ο κύριος Άσουερθ, να υπάρχει μια δυνατότητα. Είπε ότι θα το βάλει σε μια τροπολογία του ότι σε αιτιολογημένες εξαιρέσεις θα πρέπει να γίνει πιο χαλαρή η συγχρηματοδότηση. Έχουμε την έκθεση αυτή συζητήσει και στην ΚΟΝΤ. Εκεί η συγκίτρια θέλει έναν κατάλογο κρατών να καθορίσει. Αλλά αυτό δεν νομίζω πως είναι και τόσο ε, σκόπιμο αυτό, γιατί μπορεί να αλλάξουν ε, οι διαδρομές όπου υπάρχουν κάποιες δυσχέρειες, αλλάζουν οι λαθρέμποροι ε, τα δρομολογιά τους. Όπου έχετε για παράδειγμα πολύ αυστηρό ε, και εκτεταμένο έλεγχο, μια μέρα μπορεί την άλλη μέρα να είναι υπερβολικός. Θα ήθελα λοιπόν να τροποποιηθεί ενδεχομένως η κλίδα χρηματοδότησης, αλλά όχι με βάση ένα συγκεκριμένο κατάλογο. Δεν θα πρέπει εμείς να υποκαταστήσουμε τους ειδήμονες, θα πρέπει να καλέσουμε την Κομισιόν και την Όλαφ με βάση λογικά και ελέγξιμα κριτήρια να υπάρξει δυνατότητα Αύξηση της συγχρηματοδότηση, εάν είναι αναγκαίο, αλλά και αν μας το επιτρέπουν οι ε, δαπάνε του προπολογισμού. Πρέπει να έχουμε πολιτικά κριτήρια γι' αυτό. Αυτό είναι ο δικός μας ρόλος. Αλλά έναν κατάλογο κλειστό κρατών μελών δεν θα τον ενέκρινα μπορεί οποιοδήποτε κράτος μέλος από τη μια στιγμή στην άλλη να χρειαστεί και αυτό τη βοήθειά μας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σαλβαντόρ Γκαρίγκα. Δεν θα θυμόσαστε, αλλά αυτό το πρόγραμμα Hercules αφορά μια αρχική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ και πολλά χρόνια υπήρχε μια προσωρινή επιτροπή, είχε ε, συσταθεί για την παράνομη διακίνηση σιγαρέτων. Ο κύριος Μπόουμαν, ο κύριος Άσουορθ, το 1995 είχαν γίνει όλα αυτά. Τότε άρχισαν. Θα υποβληθούν τροπολογίες, Ρίτσαρτ, αλλά θα ήθελα να έχουμε λίγο περισσότερο καιρό για να δούμε το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Ο Ρίτσαρτ μιλά για αποταμίες, μάλλον για εξοικονόμηση χρημάτων από τον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην υπάρξει συγχρηματοδότηση εκεί που δεν είναι απόλυτα αναγκαίο. Ας δούμε όμως και ποιες θα είναι οι παράπλευρες συνέπειες για ορισμένες χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν μπορούν να ε, προβούν σε χρηματοδοτήση. Εκεί θα πρέπει να τονίσουμε το ε, σκέλος της συγχρηματοδότησης, γιατί έχουν μεγάλες αδυναμίες. Γι' αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε την αρχική πρόταση της Όλαφ. Δηλαδή για να εξοικονομήσουμε κοινοτικό χρήμα και απειροελάχιστες ποσότητες, δεν θα πρέπει να μην καταπολεμήσουμε τη ρίζα της κακοδαιμονίας, δηλαδή αυτή την παράνομη διακίνηση τσιγάρων, που δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στην ε, εσωτερική ένομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν ε, σοβαρές δικαιολογίες για να μειώσουμε συγχρηματοδότηση σε περιόδους που δεν θα έπρεπε καν να αγγίξουμε τη συγχρηματοδότηση, να μην την αλλάξουμε καθόλου δηλαδή. Γιάν Μούλτερ. Ευχαριστώ. Όπως και ο Σαλβαδόρ, εγώ ήμουν μέλος αυτής της πρώτης επιτροπής έρευνα το 95 που είχε συσταθεί το 95 και είχαμε υποβάλει προτάσεις που ήταν ιδιαίτερα σημαντικές που αφορούσαν και την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων διότι όλες οι πωλήσει γίνονταν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πριν ηχνηλατηθούν πέρναγε τουλάχιστον ένας χρόνος. Και θα ήθελα να πω ότι το θέμα γίνεται όλο ένα και πιο διονγκούμενο. Τη στιγμή που θεωρούμε ότι οι ήδη πόροι θα πρέπει να ενταχθούν κατά ένα συγκεκριμένο ε, τρόπο στο ε, MFF θα πρέπει να ελέγξουμε και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αλλάξουμε την ευρωπαϊκή, την κοινοτική μας μεθοδολογία. Θα πρέπει να δούμε και τους φόρους εισαγωγής. Δηλαδή να δούμε πού συλλέγονται και πού όχι σωστά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει το υψηλότερο δυνατό ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω πώς ρυθμίζεται η συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Μας ενδιαφέρει να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και τη στιγμή που υπάρχουν ήδη οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις χώρες όπου ο ΦΠΑ έχει μεγάλη σημασία, σημασία και η συλλογή γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτά. Ωραία, συνεχίζουμε αυτή τη διαλκυστίνδα. Η Ίγκια θέλει να απαντήσει. Ακριβώ για αν σκεφτεί ο καθένα το δικό του, τότε δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Θέλω να πω ότι για την συγχρηματοδότηση το μεγαλύτερο λιμάνι της Ένωσης με τη μεγαλύτερη ε, δυνατότητα εισόδου είναι το Ρότερνταμ. Πήγαμε στο Ρότερνταμ, θαυμάσιο λιμάνι. Αλλά το λιμάνι αυτό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Μέχρι τα αυτιά είναι τα λεφτά. Αν είναι κάποιο που δεν χρειάζεται επιδοτήσει, είναι το Ρότερνταμ. Και χαίρομαι που είπατε πω δεν αξιοποίησε τέτοιε πιστώσει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρή η συζήτηση, γιατί ο καθένας προσπαθεί να πέσουν στην τσέπη του από αυτό το μάνα εξ ουρανού να τον περισσότερα. Ανοίγει πολύ φαρδιά ανοιχτές στη τσέπες του. Κοιτάξτε, Γιάν, το λιμάνι του Ρότερνταμ είναι άψογο, μην ανησυχείς. Ναι, αλλά και το Αμβούργο δεν χρειάζεται επιδοτήσεις, μου φαίνεται. Για τη Μασαλία καλύτερα να μην τους δώσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ τώρα έχουμε ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Ως Επιτροπή Προϋπολογισμών βέβαια πρέπει να εξετάσουμε κυρίω σχεδόν αποκλειστικά τη δημοσιονομική πλευρά στον προπολογισμό. Αλλά πέρα από αυτήν την οικονομική πλευρά, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο συμβιώνουμε εδώ πέρα 27 διαφορετικοί λαοί σε έναν μεγάλο χώρο όπου όλα κυκλοφορούν ελεύθερα. Πολύ σημαντικός στόχος γιατί κυκλοφορούν όλα ελεύθερα και τα προϊόντα και τα πρόσωπα, τα κεφάλαια, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες και κανονισμοί ανατομέα και θέλουμε να συνεχίσει έτσι το πράγμα λόγω της επικουρικότητας, αλλά αυτό ενθαρρύνει μετακινήσεις, λάθρεμπόρια ορισμένα που θα μπορούσαν να τιμωρηθούν ποινικά, πάντως που έχουν στρεβλωτικά αποτελέσματα, ακόμα και ανθυγιεινά. Άρα η Ένωση έχει την ευθύνη να φροντίσει ό,τι βέβαια είναι παράνομο να τιμωρηθεί ή να παρεμποδιστεί και τουλάχιστον το πνεύμα του νόμου να γίνει σεβαστό είναι από τα σημαντικότερα αλλά και δυσκολότερα καθήκοντα που έχει η Ένωση και χάρη στο Κοινοβούλιο και το πρόγραμμα Ηρακλής του οποίου υπάρχουν αν κατάλαβα καλά πολλοί παρόντες εδώ από εκείνους που το σκέφτηκαν, όχι εγώ, για το λαθρεμπόριο σιγαρέτων και προϊόντων καπνού. Ο Ρίτσαρντ Άσχουερφ εξάλλου μας είπε ποιες είναι οι προτάσεις του για τον Ηρακλή 3. που ιστορικά είναι, θα έλεγα, ο 13ος άθλος του Ηρακλέους, αν θυμάμαι καλά ότι ήταν 12. Λοιπόν, για να καταλήξουμε τώρα, μήπως ο εισηγητής, ο Ηρακλής, ο τρίτος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για αυτά που είπατε τόσο πιο εύγλωτα από μένα. Έχω εντυπωσιαστεί από μερικά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, από τις ενθυμίσεις τους δηλαδή από το 1995 και την εμπειρία τους. Εγώ δεν είμαι τόσο παλαιός βουλευτής, αλλά θα τα λάβω όλα αυτά υπόψη μου. Τέλος πάντων, τα σοβαρά είναι ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Γκάις ότι πρέπει να επιδείξουμε πνεύμα ευθύνης εδώ. Πολύ σοβαρά τα παίρνω υπόψη μου αυτά τα σχόλια, αλλά απ' την άλλη πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα και εδώ με ενθαρρύνουν πολύ αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλε. Αλλά παραμένω ανοιχτός σε προτάσεις και συστάσεις των συναδέλφων και θα συνεχίσω να τους διαβουλεύομαι, να τους συμβουλεύω. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. η Γιούτα και ο Σαλβαδόρ μου έλεγαν ότι στην Επιτροπή όταν προείδρευε η κυρία Τεάτο όχι, προείδρευε της Επιτροπής Κόντ και ο εισηγητής τότε ήταν, λέει ο Σαλβαδόρ, ένας συντηρητικός, Άγγλος συντηρητικός, ο κύριος Μπόμαν. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη συντηρητική παράδοση σε αυτά τα θέματα. Αλλά θα υπάρχουν και τροπολογίες από άλλες ομάδες βέβαια. Λοιπόν, για το χρονοδιάγραμμα, για τη συνέχεια. Η διορία κατάθεση τροπολογιών λύγει στις 15 Οκτωβρίου. Θα ψηφίσουμε την έκθεση του Ρίτσαρντ στις 6 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή Κόντ στις 15 και θα, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου θα περάσει. Αυτά συνάδελφοι, ευχαριστούμε και τον εισηγητή. Έληξε η ημερήσια διάταξη. Κερδίσαμε χρόνο λοιπόν διότι δεν χρειάζεται να συνεδριάσουμε το απόγευμα αλλά και ούτε και στη συνέχεια του πρωινού. Στο ίδιο πνεύμα πριν φύγουμε θα ήθελα να σας προτείνω κάτι για την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα μερικοί θα έχουν πάρα πολλή δουλειά σε σχέση με τον προϋπολογισμό διότι έχουμε το πρόγευμα με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 τον τριμερή διάλογο ή μάλλον την ομάδα επαφής το πρωί και το προετοιμασία του τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό 13. Και έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής μας όλη την 5η 18. Μετά από διαβούλευση με τη γραμματεία και όλα όσα κάναμε χθες και σήμερα σας προτείνω να γίνει η συνεδρίαση της Πέμπτης μόνο το πρωί. Αν συμφωνείτε προβλέψαμε συνεδρίαση των συντονιστών στις 2. Μα την κρατήσουμε προς στιγμή αυτή τη δυνατότητα για τους συντονιστές και συντονίστριες να δούμε αν τη χρειαζόμαστε. Αλλά πάντως μπορούμε ήδη να πούμε ότι το απόγευμα της 5ης 18 δεν χρειάζεται να συνδυάσουμε εκτός αν κανείς επιμένει απόλυτα να εργασθώμεν το απόγευμα της η Συμφωνείτε. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει Σαλβαδόρ. Την 5η 18 το πρωί. Πρωί. Σας αφήνω να πάτε στο Βουκουρέστι. Τι άλλο να σας κάνω. Δεν μπορώ να καταργήσω τελείως τη συνεδρίαση. Ο Σαλβαδόρ είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΕΛΚ. Οπότε πρέπει να είναι στο Βουκουρέστι. Λοιπόν, έτσι θα πράξουμε λοιπόν λίγη συνεδρίαση. να μην ξεχάσετε τις κάρτες σας να τις ξαναπάρετε.